Δύναμη Δυνάμει του άρθρου 149 του κανονισμού, το Προεδρείο ενέκρινε το τελικό σχέδιο μερίσιας διάταξης, το οποίο έχει και διανεμηθεί. Σε συμφωνία με τις ομάδες προτείνω τις εξής αλλαγές στο σχέδιο μερίσιας διάταξης. Μετά την ώρα των ψηφοφοριών θα γίνουν δηλώσεις από το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τις συνέπειες της, απόφαση απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με την απόφαση ασφαλούς για τις, των Ηνωμένων Πολιτειών, σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η Επιτροπή των Οικονομικών Υποθέσεων έκανε δεκτές δύο εκθέσεις για το ΕΕΣΥ Οικονομικό ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Επενδύσεις και την προκήρυξη των θέσεων ε, Διευθυντού Διευθυντρίας. Θα ψηφιστεί αυτό στη σημερινή ψηφοφορία και ως εκ τούτου παρατείνεται η συνεδρίαση ω τις 11. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Με τι ε, τροποποίησεις αυτές λοιπόν εγκρίνεται. Η Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων εξέτασε τις, ε, την έκθεση ασυλίας για τον κύριο Σπιεύκα που θα ψηφιστεί κατά τη διάρκεια των σημερινών ψηφοφοριών. Και έχω λάβει τα έξι αιτήματα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ζητεί η συζήτηση σχετική με τι δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για τι συνέπειε τη αποφάση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για, το ασφαλές, για τον ασφαλή λιμένα ΗΠΑ να ψηφιστεί ολοκληρωνόμενη από ένα ψήφισμα κατά, το τρίτο, κατά την τρίτη περίοδο συνόδου, Σύνοδου της, ε, του Οκτωβρίου. Κονσάλης Πόνς, παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο, κύριος Γκονσάλης Πόνς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, ε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ζητά η συζήτηση που θα έχουμε το απόγευμα ε, για την απόφαση για, το, για τον ασφαλή λιμένα να συμπληρωθεί από ένα ψήφισμα, γιατί διαπιστώσαμε ότι τα δεδομένα των συμπολιτών μας και των επιχειρήσεών μας δεν είναι τόσο ασφαλή όσο πιστεύαμε. Θα θέλαμε λοιπόν το συντομότερο δυνατό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάρα αυτά γίνεται, να θεσπίσει μια πρόταση για να ξεφύγουμε από αυτό το νομικό κενό στο οποίο βρισκόμαστε εξαιτίας αυτής της απόφασης ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ευχαριστώ. Κύριε Κονσάλε Πόνς, προβλέπετε η συζήτηση. Υπάρχει δήλωση Συμβουλίου και Επιτροπής. Το ζήτημά μας είναι τώρα το ψήφισμα. Το έτοιμά σας δηλαδή αφορά μόνο το αν επιπροσθέτως θα υπάρξει ψήφισμα για την προσεχή περίοδο συνόδου στο Στρασβούργο που θα ψηφιστεί. Ε, θέλει κανείς να υποστηρίξει το αίτημα η κυρία Χολμάιερ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συμφωνούμε νομίζω ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αγκυρώνει τη συμφωνία περί ασφαλούς λιμένος είναι πάρα πολύ σημαντική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λόγω των πιέσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ιδιαίτερως μαζί με άλλες ε, ομάδες ε, δείχνει ότι ήταν ανεπαρκής αυτή η συμφωνία. Δεν υπάρχει επαρκής προστασία δηλαδή από τη συμφωνία αυτή και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να συνεχίσει τις προσπάθειες με ένα ψήφισμα που θα εγκρίνουμε από κοινού για να τοποθετηθούμε αφενός, αφετέρου δε για να προχωρήσουμε ταχύτατα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αναζήτηση ενός τρόπου με τον οποίο μπορούμε να ρυθμίσουμε το ζήτημα της ε, διαβίβασης πληροφοριών, ε, δεδομένων μάλλον από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ΗΠΑ και Τούμπαλιν. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς να ταχθεί κατά τις προτάσεις, παρακαλώ. Κυρία Ζήπελ. Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντική αυτή η απόφαση και χαίρομαι που ακούω από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αυτά τα λόγια, γιατί εγώ είχα ακούσει άλλου είδους τοποθετήσεις από αυτή την πλευρά. Για το ψήφισμα. Το, το Κοινοβούλιο χρόνια τώρα έχει σαφή θέση σε σχέση με το Safe Harbor, ότι δηλαδή δεν είναι ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα με την συμφωνία αυτή. Και δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε για άλλη μια φορά. Η μπάλα βρίσκεται πια στο γήπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή πρέπει να μας πει πώς θα αντιμετωπίσει το ζήτημα. Δεν μπορεί δηλαδή να συνεχίσει να πράττει όπως έπρεπε μέχρι τώρα. Πρέπει να κάνει συγκεκριμένε προτάσεις και πάνω σε αυτές θα πρέπει να αντιδράσουμε εμείς. Ο Πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, καλώς ψηφίζουμε την πρόταση του κύριου Κονσάλης Παρακαλώ, διανατάσεως. Κατά. Απερίφθη νομίζω. Πολύ καλά. Αρχίζει λοιπόν η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν οι πάντες. Ξαναρωτάω. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Η ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς έχει καταθέσει έτοιμο για δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και είπα της εκπροσώπου για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με την κατάσταση στην Τουρκία μαζική φόνη αθώων σε ειρηνική διαδήλωση και δίνω το λόγο για το θέμα αυτό στον κύριο Χατζηγεωργίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήταν μεγάλο λάθος αυτής της ολομέλειας να δει αυτό το θέμα ως μια άλλη επίθεση αυτοκτονίας. Η εκατόμβη των νεκρών μας υποχρεώνει να δούμε προς τα που οδεύει η χώρα αυτή μετά από το αίμα τόσων νεκρών αλλά και με τόσους άλλους νεκρούς τους τελευταίους μήνες μεταξύ των τουρκικών δυνάμεων και των Κούρδων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να συζητήσει το θέμα αυτό σε βάθος, εκτάκτος και σήμερα. Δεν παίρνω τον λόγο ως κάποιο που θέλει να αδικήσει την Τουρκία Αντίθετα, θα έχουμε όλοι όφελο από μια έγκαιρη και σε βάθο συζήτηση του ζητήματο. Η διχόνοια που ελοχεύει στη χώρα μπορεί να τη σπρώξει προ το χάο και εμεί πρέπει να αντιστρατευτούμε αυτή την πορεία. Η έκφραση αλληλεγγύη προ του Τούρκου πολίτε και η ενό λεπτού σιγή που δεν έχουμε κάνει δεν πρέπει να αποτελεί άλοθη για να αποφύγουμε μια ολοκληρωμένη συζήτηση. Στόχος μας πρέπει να είναι να αποφύγουμε μετά τον αραβικό χειμώνα τον πιθανό τουρκικό χειμώνα. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θέλει κανείς να υποστηρίξει το αίτημα. Θέλει κανείς να προβάλλει αντιρρήσεις. Όχι, ψηφίζουμε λοιπόν. Υπέρ παρακαλώ, για να Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Και παίρνω στο επόμενο θέμα της σημερινής της διάταξης που είναι η προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15 και 16 Οκτωβρίου.